σήμερα με βάση το άρθρο 231.4 ε, των διορθωτικών ε, ε εγκρίνονται ε, τα πρακτικά, τα διορθωτικά πρακτικά των αρμοδίων επιτροπών. Ε, υπάρχουν στην δικτυακή, στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας.